στο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτή την ανησυχία μας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Δαμανάκη. Η συζήτηση για την κατάσταση στο Ιράν λοιπόν ολοκληρώθηκε και θα ψηφίσουμε μετά την εξέταση του της επόμενης συζήτησής μας που είναι η Αίγυπτος. Και συγκεκριμένα η υπόθεση του blogger αλλά Αμπτέλ Φατά. Ο κύριος Καμίνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε παρακολουθήσει με πολλές ελπίδες και καλωσορίσαμε αυτά που έγιναν την Άνοιξη στην Αίγυπτο. Ε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε μια χώρα με πάνω από 70 εκατομμύρια κατοίκους και μια, ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτισμό για όλο τον αραβικό κόσμο. Και γι' αυτό ε, θεωρούσαμε ότι η Αίγυπτος είναι ένα παράδειγμα δημοκρατικής αλλαγής. Και θέλαμε βέβαια η Αίγυπτος να είναι παραδειγματική χώρα όσον αφορά τον εξοχρονισμό και την δημοκρατική τη λειτουργία μέσα στα πλαίσια του Ισλαμικού κόσμου. Θα θέλαμε να μπορούμε να πούμε ότι οι αραβικές, Ισλαμικές χώρες ε, ε, ασπάζονται τις δημοκρατικές ε, αξίες που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Δυστυχώ έχουμε όσο πάει και περισσότερα μηνύματα που καταδεικνύουν ότι είναι ανασυχητικά αυτά που διαμείβονται στην Αίγυπτο σήμερα. Έχουμε πολλές ε, περιπτώσεις ε, καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως παραδείγματο χάρη τα δικαιώματα των κόπτων χριστιανών στην Αίγυπτο που βλέπουν ε, συνεχώς να καταπατούν τα δικαιώματά τους. Και επίσης αυτό που έχουμε τώρα με την ελευθερία του λόγου. Θα πρέπει λοιπόν να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα στο λαό, στην κυβέρνηση της Αιγύπτου, ότι χαιρετίζουμε τις αλλαγές που έλαβε η χώρα, αλλά θέλαμε να είναι θετικές και ειρηνικές. Το Γεγονό ότι ο Μουμπάρακ εγκατέλειψε την θέση του Προεδρού άνοιξε το δρόμο για μια μεταβατική κυβέρνηση στην Αίγυπτο. κατά τη διάρκεια μιας ε, ειρηνικής διαδικασίας υπέρ των δικαιωμάτων των χριστιανών κοπτών της Αιγύπτου οδήγησε σε ε, πολλούς ε, θανάτους και πάνω από 300 τραυματίες. Αυτό φαίνεται ότι οι Αιγυπτιακές αρχές έχουν χάσει το μέτρο σε ό,τι αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Η μοίρα μάλιστα του Αλά Αμπτελ Φατάχ, του μπλόγκερ αυτού, καθώς επίσης και πολλών άλλων χιλιάδων Αιγύπτιων των ε, πολιτών ε, δείχνει ότι οι Αιγυπτιακές αρχές ε, χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή αυταρχικές μεθόδους. γίνεται ταυτόχρονα παραβίαση και του άρθρου 10 της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρέπει να πιέσουμε την προσωρινή κυβέρνηση να επιστρέψει στη χρήση πολιτισμένων μέσων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε πολλοί εδώ πέρα που χαιρετήσαμε την Αραβική Άνοιξη, αλλά η επανάσταση δεν παίρνει τον ίδιο δρόμο παντού. Οι Τινήσοι ακολουθούν ένα δημοκρατικό πλαίσιο ε, που κανένας δεν αμφισβήτησε. Δυστυχώς όμως είναι η μόνη χώρα για την οποία μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Στη Λιβύη γίνεται λόγος να καθιδρυθεί η Σαρία. Στην Αίγυπτο, ε, στη Συρία πολλές ε, δολοφονίες, γίνονται πολλές δολοφονίες και η κατάσταση στην Αίγυπτο επίσης μας ανησυχεί. Στις 30 Οκτωβρίου ε, ο Αλά Αμπτέλ Φατά, blogger, συνελήφθη. Και η σύντροφός του το ίδιο. Και οι δύο αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τα στρατοδικεία είναι σύμβολα του Αιγυπτιακού λαού, σύμβολα αντίστασης ε, και αγώνα για την ελευθερία. Ε, ακόμα και σήμερα κριτικάρουν το καθεστώ και του ε, στρατιωτικού. Χωρί ελευθερία σκέψη και έκφραση δεν είναι δυνατόν να εγκαθιδρυθεί μια δημοκρατία. Δέκα μέρε πριν από τι εκλογέ στην Αίγυπτο πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προ τι Αιγυπτιακέ αρχέ, έτσι ώστε να εγγυηθούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα όλων των πολιτών του. Ευχαριστώ. Now, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βεϊτζενίν τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε συγκεκριμένες υποθέσεις ε, του μπλόκερ ε, Αλάμπτελ Φατάχ και του συναδέλφου του ε, Σανάντ. Εμείς απαιτούμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, αυτές οι υποθέσεις είναι συμπτώματα μιας κατάστασης. Ε, που επικρατεί στην Αίγυπτο. Έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες για την ε, καταπίεση των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους, τους δημοσιογράφους. Πάνω από 12.000 πολίτες δικάστηκαν από στρατοδική από το Μάρτιο μέχρι τώρα. Ε, ακόμα ισχύει το στρατιωτικό κράτος, στρατιωτικό καθεστώς ε, δεν ξέρουμε ακριβώς ε, τι συμβαίνει στο Κάιρο. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι ε, Αιγυπτικές αρχές οφείλουν πολλά στον ίδιο του το λαό και σε εμάς τους Ευρωπαίους που ελπίζουμε για καλύτερο μέλλον για την Αίγυπτο. Ξέρουμε από τη δική μας ιστορία ότι ο δρόμος για τη δημοκρατία είναι περίπλοκος, δύσκολος και μακρύς αλλαγή ε, του Μουμπάρακ, η φυγή του Μουμπάρακ ε, σίγουρα ήταν ένας, μια τεράστια σεισμική δόνηση με πολλούς μετασυσμούς. Όμως θέλουμε να είμαστε βέβαιοι για την κατεύθυνση προς την οποία θα κατευθυνθεί η Αίγυπτος, ότι αυτή η πορεία που ξεκίνησε θα συνεχιστεί και ότι θα είναι ένας δρόμος προς τη δημοκρατία, σταθερός. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η κυρία είναι Πρέπει να υποστηρίξουμε τον λαό της Αιγύπτου στον αγώνα του για δημοκρατία. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, στην ε, διάμεση μεταβατική αυτή περίοδο, ε, σε διεθνές επίπεδο να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την, ε, ε της παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με αυτό μας το ψήφισμα θέλουμε να κάνουμε μια έκκληση προς το στρατιωτικό καθεστώς υπέρ του blogger Αλά Αμπτέλ Φατά, του οποίου περίπτωση όπως και πολλές άλλες ε, κρίθηκε ενώπιον στρατιωτικού δικαστηρίου, στρατοδικίου δηλαδή. Ε, γνωρίζετε επίσης ε, ότι ο στρατός ε, κατέπνιξε μια πυρηνική διαδήλωση στο Μαρινάπ και αυτό οδήγησε στο θάνατο δεκάδων πολιτών και τον τραυματισμό εκατοντάδων. Θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο Αιγυπτιακό καθεστώς έτσι ώστε να κάνει σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Thank you, President, Commissioner, colleagues. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Η νέοι, γέροι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έχουν μιλήσει καθαρά. Θέλουν το δικό τους μέλλον, ευκαιρίες, ε, να πάψει η διαφθορά, θέλουν να γίνουν σεβαστά η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συρίζουμε αυτό το αίτημά τους για ελευθερία και είμαστε ταπεινοί σε σχέση με αποφάσεις που έλαβαν στο παρελθόν ε, διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά είμαστε και προσιλωμένοι στη δημιουργία μιας εγκρινήσιας συνεργασίας με την Αίγυπτο στο μέλλον. Μα με ποια Αίγυπτο. Ελπίζω πως θα μπορούμε, δεν να μιλήσουμε για μια νέα Αίγυπτο, αλλά βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο δείχνει τα ίδια χαρακτηριστικά και τι ίδιε συμπεριφορέ όπω ο Χώστη Μουμπάρακ. Ανησυχώ. Πάνω από 12.000 πολίτε δικάστηκαν από τα στρατοδικεία από την ε, Επανάσταση και μετά. Αυτή η αδικία θα πρέπει να πάψει. Είναι πέρα αυτών των Αιγυπτίων που πιστεύουν πω τα στρατοδικεία δεν είναι νόμιμα. Ε, δεν, και αυτό ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 10 της Καθολικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο εκτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλά Αμπτέλ Φατάχ είναι ένα ακόμα θύμα. Αύριο θα γιορτάσει τα γενέθλιά του. Γίνεται 21 χρονών μέσα σε μια φυλακή υποφρικτές συνθήκες. Περιμένει να ε, καταπέσουν οι κατηγορίες εναντίον του. Επίσης περιμένει να γεννηθεί το πρώτος του γιος. Η γυναίκα του ε, ε, είναι ετοιμόγενη. Επίσης είχαν ελπίδες για μια νέα γενιά, μια νέα ευκαιρία. Ο γιος του θα ονομαστεί Χαλέντ, στο προστιμήν του Χαλέντ Σαΐτ που δολοφονήθηκε από την αστυνομία. Ο Ελφατάχ είναι ένα σύμβολο. Σύμβολο είναι και πολλοί άλλοι που έχουν βασανιστεί στη χώρα αυτή. Η ειρηνική πορεία της Αιγύπτου προς τη δημοκρατία θα πρέπει να γίνει μέχρι της απελευθέρωσης των πολιτών και των πολιτικών κρατουμένων, καθώς και των κρατουμένων συνείδησης, των αντιρρησιών συνείδησης. Νομίζω πως θα έπρεπε αυτό το ψήφισμα εξαιρετικά να μεταφραστεί και στα αραβικά καθώς και ότι το όνομα του κυρίου Αλάχ Αμπτελ Φατάχ είναι λάθος γραμμένο στο ψήφισμα και πρέπει να διορθωθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπραντνερ. Ε, στην Αίγυπτο δεν έχουμε μόνο νέα πρόσωπα. Ε, 28 Νοεμβρίου οι εκλογέ ε, πλησιάζουν και όσο πάει υπάρχουν περισσότερε απελίε κατά ατόμων. Το Μάτι του 2011 πάνω από 12.000 ε, ε, άτομα έχουν δικαστεί από στρατοδικεία. Πολλοί όπως ο, αλλά Αμπτελφάραχ έχουν ε, βασανιστεί, περιμένουν στις φυλακές. Η ατμόσφαιρα, το περιβάλλον στην Αιγύπτο δεν προωθούν την, ε, ε, οργάνωση δημοκρατικών εκλογών. Ακούμε πολλά κενά λόγια και φαίνεται ότι η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι τόσο καλή. Η κυρία Άστον σε μια επιστολή της του 28 Οκτωβρίου ε, καλεί την Αίγυπτο να υιοθετήσει τα απαραίτητα βήματα προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει η Αίγυπτος επιτέλους να εφαρμόσει τις υποσχέσεις της. Όπως είναι αλφα σοκ που μίλησε προηγουμένως, ζητήσαμε από τον είπα εκπρόσωπο να ξαναεξετάσει το θέμα, να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει πλειστά καταδικάσει την ε, ε, στάση του, της Αιγύπτου θα πρέπει να μην χάσουμε τη μικρή αξιοπιστία που έχουμε ακόμα στην περιοχή με τις στάσιμες. Θα πρέπει να προωθήσουμε την σοβαρή λήψη υπόψη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία. Μπορεί να είναι, μπορούν να είναι περήφανοι οι Αιγύπτιοι για αυτό που έχουν πετύχει θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να πετύχουν τις ελπίδες και τα όνειρά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πράντνερ. Περνάμε στου εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, κυρία Μακοβέη, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ο blogger Αλά Αμπτελ Φατά είναι ένας από τους 1200 περίπου πολίτες που έχουν δικαστεί από στρατοδική από την αρχή της Επανάστασης στην Αίγυπτο συνελήφθη κατόπιν μιας ειρηνικής διαδήλωσης ε, χριστιανών κοπτών στις 9 Οκτωβρίου που οδήγησε στην πιο βίαιη αντίδραση των, ε, ε, των αρχών της Αιγύπτου μετά από την πτώση του Μουμπάρακ. βρήκαν το θάνατο 25 άτομα ενώ 300 ακόμα τραυματίστηκαν. Τόσο η Κομισιόν όσο και το Συμβούλιο πρέπει να απαιτήσουν από τις Αιγυπτιακές αρχές να θέσουν τέρμα στις ε, δίκες πολιτών από στρατοδικεία και ταυτόχρονα θα πρέπει να απελευθερώσουν όλους αυτούς τους πολιτικούς ε, ε, ε, κρατούμενους και κρατούμενους συνείδησης. Θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη και αντικειμενική έρευνα, διερεύνηση των γεγονότων που ακολούθησαν την ειρηνική διαδήλωση της 9 Οκτωβρίου των κοπτών χριστιανών. Θα πρέπει όλοι μαζί να μεριμνήσουμε έτσι ώστε η επανάσταση να οδηγήσει σε μια πραγματική δημοκρατία. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέρινγκ και Όντενμπεργκ, μέρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η φυλάκιση του Αλα Αμπτελφατά ε, είναι ένα ανησυχητικό παράδειγμα της ε, ε, χειροτέρευσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Ο Αλά Αμπτελ Φατάχ ήταν ένας ε, πραγματικά πολύ καλός δημοσιογράφος που περιέγραψε πολύ καλά το τι συνέβη στις 9 Οκτωβρίου στην Αίγυπτο. Ε, οι στρατιωτικοί μετά από αυτά τα γεγονότα τον ε, κάλεσαν να να δικαστεί. Αυτός αρνήθηκε να δικαστεί από στρατιωτικό και γι' αυτό κρατείται. Η περίπτωση του βέβαια δεν είναι μοναδική. Η ε, προσωρινή κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να ε, προσάγει και να φυλακίζει τόσο ειρηνικούς διαδηλωτές όσο και τους δικηγόρους τους. Πάνω από 1.200 άτομα έχουν συλληφθεί από το Μάρτιο και μετά. τα δικαιώματα ελευθερίας έκφρασης και γνώμης θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Αλάχ αβδελφατάχ Φατάχ είναι ένας άνθρωπος ε, του ίντερνετ ήδη συνελήφθη τον καιρό του Μουμπάρακ γιατί ε, είχε φτιάξει διάφορα blog τα οποία λειτουργούσαν τον καιρό της δικτατορίας. Η σύζυγός του δε, δε είπε πως δεν υπήρχε λόγος να γυρίσουν προς τα πίσω και εκείνοι ε, δημιούργησαν μαζί ένα blog αντιπολίτευσης που είναι από τα πιο αναγνώσιμα στην Αίγυπτο επέστρεψαν στην Αίγυπτο λοιπόν, ήταν στην ε, πλατεία Τεχρήρ και, με, και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Και έπειτα μετά από την Επανάσταση ε, συνέχισαν να υπαγρυπνούν με τον ίδιο τρόπο όπως και στο καθεστώς του Μουμπάρακ. Και αυτό τους τύχησε τη φυλάκιση με κατηγορίες ε, τελείως ε, ε αστήρικτες. Η αδερφή του, η κυρία Ισαΐφ, που είναι μέλος εμ επίσης έχει συλληφθεί μέσω από δίκηση στρατοδικείο είναι ακόμα ένα άνθρωπος, ακόμα μία γυναίκα της Αιγύπτου που είναι αξιοθαύμαστη γιατί συνεχίζει να αγωνίζεται. Εμεί εδώ λέμε πως τους θυμόμαστε και πως είμαστε στο πλευρό τους, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι ακόμα. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ευάρες και με αυτό το νέο στρατιωτικό καθεστώς. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει άλλο ένα καθεστώς ε, Μουμπάρακ χωρίς το Μουμπάρακ. Δεν πρέπει να είμαστε καθόλου καθόλου μαζί τους. Υπήρξαν κατηγορίες ε, ε, μη ανοχής σε θρησκευτικά θέματα. Είμαστε Ε, γίνεται μια διαδικασία που προσπαθούν να βρουν ε, οι ε, συμμαχίες για να προστατεύσουν τις μειονότητες. Εμείς πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή όμως για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή πρέπει να είναι η στάση μας από εδώ και μπρο. Ο κύριος Τζαρνέσκι. Obserwujemy regres, obserwujemy cofanie się, gdy chodzi o Πρόεδρε, ε, βλέπουμε να υπάρχει μια υπεναχώρηση όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Η δημοκρατία αυτή του λαού που επρόκειτο να φέρει ανθρώπινα πρότυπα είναι ουτοπία φαίνεται. Αυτό που μας πριν από αρκετούς μήνες ότι δεν αρκεί να φύγουν οι δικτάτορες, αλλά ότι πρέπει επίσης να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από τους δικτάτορες, ποιοι αναλαμβάνουν την ισχύ. Αυτοί που μας προειδοποίησαν έτσι, φαίνεται, είχαν δίκιο τελικά. Υπήρχε αυτή η ουτοπία ε, ελευθερίας που σήμερα έχει εξαφανιστεί και όσον αφορά την ελευθερία του λόγου εγώ το λέω αυτό που είμαι και εγώ blogger εδώ και 7 χρόνια και γι' αυτό είμαι απόλυτα αλέγγυος με εκείνους που διώκονται στην Αίγυπτο. Κύριος Μαστάλκα, η περίπτωση Αλα Αμπτελ Φατάχ είναι ένα μόνο παράδειγμα της αδυναμίας των δικών μας πολιτικών η περίφημη, η περιβόητη άνοιξη, αραβική άνοιξη ε, τελειώνει με ε, καταπίεση των ανθρώπων που ε, εκφράζουν την αντίδρασή τους. Ε, δεν πρέπει να συμπλέουμε με ανθρώπους που είναι απλώς ε, κυνηγούν απλώς την εξουσία ε, φωνάζοντας δημοκρατικά σλόγγαν. Οι γρήγορες ε, λύσεις οδηγούν σε νέα και περισσότερα προβλήματα μόνον. Ε, και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αυτό που είδαμε και πριν τον πόλεμο του Ιράκ. Πολιτική σύγκρουση με το Ιράκ με το Ιράν ε, χωρίς ε, προσπάθειες ε, έβρεσης μιας ενός ενδιάμεσου δρόμου. Ε, είναι εύκολο να είμαστε πολεμοχαρείς. Είναι δύσκολο να βρίσκουμε συμβιβασμούς. Η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό καθήκον είναι να επιβάλλει τα δημοκρατικά ιδεώδη ειρηνικά. Καταλαβαίνω ε, πώς είναι δυνατόν να ε, ε δεχόμαστε την είσοδο τουρκικού στρατού στη Συρία για την, καταπο, για την καταπολέμηση των Κούρδων και να μην δεχόμαστε το ίδιο από τη Συρία, Συριακό καθεστώς, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Η Αίγυπτος είναι μια πολύ ωραία χώρα, πολύ όμορφη και με ρομαντικό, ρομαντική ιστορία όμως οι δραστηριότητες της στρατιωτικής χούντας δεν τις έκαναν καμία χάρη, δεν την εξυπηρέτησαν και το να επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη και το λέω αυτό ως χριστιανός εγώ ίδιος και μέλος του ΕΛΚ που είναι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να στηρίξουμε τους χριστιανούς και όλους ε, όσους ε, υποφέρουν λόγω θρησκείας στον κόσμο. Η περίπτωση του κυρίου Φάταχ είναι πολύ σημαντική σήμερα. Πρέπει να το συγχαρούμε για το θάρρος του που δεν δέχτηκε την ε, κατάσταση και δεν ε, μείωσε την επαγρύπνησή του. Επίσης, Πρέπει να στηρίξουμε το κίνημα που ζητά από όλους τους Αιγυπτίους να μην στηρίξουν την, το, στρατιωτική, το στρατιωτικό καθεστώς που επικρατεί αυτή τη στιγμή και έτσι θα εξυπηρετήσουμε ολόκληρο το λαό της Αιγύπτου. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Η κυρία Κρέτου. Κύριε Πίτροπε, όλοι χειροκροτήσαμε τις αλλαγές της ε, Αραβικής Άνοιξης. Ε, ήμασταν όλοι πέρα των όσων αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία στο κέντρο του Καΐρου. Ο δυστυχώς όμως ε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η δημοκρατία δεν έχει επικρατήσει. Το στρατός καλά κρατεί και αγνοεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Ε, μάλιστα, ε, οι διάφορες μειονότητες έχουν δεχτεί επιθέσεις όπως η μειονότητα των κοπτών. Πάνω από 12.000 πολίτες δικάστηκαν από στρατοδικία μετά από την πτώση του καθεστώτος του Μουμπάρακ, πράγμα το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά όσον αφορά τη βιωσιμότητα αυτής της ε, διαδικασίας εκδημοκρατισμού. Ο κύριος Ελφατάχα βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Αρνήθηκε να περάσει το που θεωρεί ότι δεν είναι αμερό και εγώ συμφωνώ με όλους όσους ζήτησαν την απελευθέρωση του Αλλάχ Αμπτελ και ζητάμε επίσης να γίνει μια δίκαιη δίκη ενώπιον ενός πολιτικού δικαστηρίου με σεβασμό του δικαίου. Πρέπει πιο πολύ να προσέξουμε τα όσα συμβαίνουν στην Αίγυπτο για να μην ξαναγίνουν τέτοιου είδους παραβιάσεις. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κορχόλα είναι η επόμενη ομιλήτρια στο Κάιρο στις 9 Οκτωβρίου 25 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατόπιν της ε, δράσης της επέμβασης του στρατού ε, κατά τη διάρκεια μιας ελληνικής διαδήλωσης. Ε, και άλλοι τέτοιου τύπου γεγονότα έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους μήνες. 12.000 άτομα έχουν δικαστεί από στρατοδικία τα τους τελευταίους μήνες. Η περίπτωση Αλα Αμπτελ Φατάχ είναι ενδεικτική και εμβληματική. Ο Αμπτέλ Φατάχ αρνήθηκε να δικαστεί από, από τα στρατοδικεία, ήταν, αυτό ήταν πολύ γενναίο, αλλά τον οδήγησε στη φυλακή. Η κατάσταση στην ε, Αίγυπτο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, διότι η Αίγυπτος ε, ζει μια μεταβατική περίοδο. Ο τύπος ε, και οι δημοσιογράφοι έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να τους προστατεύσουμε θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να μην είναι ανοιχτή η πολιτική οδό στην Αίγυπτο και να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίε και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε όσου αγωνίζονται για αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητήσαμε στην περασμένη ορομέλη για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Το θέμα ξανά ήρθε μπροστά μας. Επιτροπός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν ότι η μείωση του χώρου ελευθερίας στην Αίγυπτο έχει μειωθεί. Εγώ είμαι με το μέρος εκείνο που ζήτησαν άμεση απελευθέρωση του Αμπτελ Φατά, ενός blogger που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή επειδή είναι αντίθετος με το καθεστώς. καταδικαστεί από το δικείο γιατί τόνισε να επικρίνει τις δράσεις των δυνάμεων ασφαλείας ε, κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Ο Μπτέλφαντα έγραφε από το ε, κελί 19 στη φυλακή και ε, έλεγε εντάξει εγώ δεν περίμενα να ξαναβρωθώ στη φυλακή μετά την επανάσταση στην Αίγυπτο. Όπως είπαν ήδη οι συνάδελφοι, θεωρώ ότι οι φυλακίσεις και οι δίκες κατά των ατόμων αυτών σε στρατοδικία πρέπει να σταματήσουν. Δεν πρόκειται η δημοκρατία. Ευχαριστώ λοιπόν. Θα περάσουμε στο ΚΑΣΔΙ. Η κυρία Ζαμπόρσκα βλέπω έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο blogger Abdul έχει κατηγορηθεί ότι κινητοποιεί κατά των ε, στρατιωτικών δυνάμεων ε, μέσα στα πλαίσια των ε, διαδηλώσεων και κατηγορείται ενώπιον στρατιωτικού παρόλο που δεν ήταν στρατιώτης. Πολλοί από αυτούς που είναι εκείνοι που πρόθεσαν την βία εξακολουθούν να βρίσκονται ελεύθεροι. Ξέρουμε, στη Σλοβακία είχαμε παρόμοια κατάσταση το 88 στη Ζιμπρατισλάβα. Οι κομμουνιστές ε, χρησιμοποίησαν μια παρόμοια στάση. Χριστιανοί που ζητούσαν τον σεβασμό των βασικών τους δικαιωμάτων διώχθησαν. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος όλων των χριστιανών αποστείλει ένα σαφές μήνυμα προς την Αίγυπτο ούτως ώστε οι Αιγύπτιοι να κατανοήσουν ότι η Ευρώπη ζητά το σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικά την ελευθερία του λόγου. Θα πρέπει να εγγυηθούν αυτά τα δικαιώματα, αλλιώ δεν υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα αυτή. Ο η κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη ε, και γενικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, έχουν ε, βοηθήσει να τηρείται ενήμερη κοινωνία. Χωρίς αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη Συρία για παράδειγμα, δεν θα ξέραμε τι συμβαίνει. Χιλιάδες άτομα διακινδυνεύουν τη ζωή τους τοποθετώντας πληροφορίες στο ίντερνετ και εμείς μαθαίνουμε τι συμβαίνει στη Συρία με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τη δημοκρατία η ενημέρωση, ε, η ελευθερία της ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Ο Αλά Αμπτελ Φατάχ βρίσκεται κρατούμενος θύμα της ε, δράσης των στρατιωτικών αρχών της Αιγύπτου. Ε, και αυτό εξαιτία του μπλοκ του. Σίγουρα αν δεν τηρούσε αυτό το μπλοκ δεν θα είχε και τα συγκεκριμένα προβλήματα. Η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία γνώμης είναι θεμελιώδες δικαίωμα δεν μπορούμε να επιτρέπουμε παραβίασή του. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αυταρχισμό στην Αίγυπτο με δημοκρατικά μέσα. Είναι κρίμα που μετά την, Αιγυπτιακή, την ε, Αραβική Άνοιξη έχουμε φτάσει το φθινόπορο των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι χριστιανοί υφίστανται ε, μαζικές ε, ε, πιέσεις ε, και δεν τους υποστηρίζουμε αρκετά θα πρέπει σε παρόμοιες περιπτώσεις ε, με επιθέσεις εναντίον χριστιανών οπουδήποτε στον κόσμο να αντιδρούμε αμέσως ε, και ιδιαίτερα βέβαια αυτό αφορά την Αίγυπτο. Ε, καταδικάζουμε τις δράσεις, τις πράξεις αυτές και ζητούμε από την Αίγυπτο να διορθώσει την κατάσταση. Κύριε Σας ευχαριστώ. Κύριε Καραστερή, το λόγο μετά ή είναι μπλε κάρτα που έχετε δείξει. Α, μετά. în cazul Αν συγκρίνουμε το Αιγυπτιακό καθεστώς με τα καθεστώτα που αγνοούν τις ανθρώπινα δικαιώματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το, η κατάσταση του Αλά Φατάχ δεν θα ήταν τόσο σοβαρή, όμως η Αίγυπτος θέλει να γίνει δημοκρατική και πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνονται σεβαστά. Σε μια πραγματική δημοκρατία οι πολίτες δεν δικάζονται από στρατοδικείο. Αυτό μπορεί να φαίνεται κάτι που είναι ίσονο σημασία, αλλά δεν είναι. Τέτοιου ε, καταστάσεις μπορεί να ανοίξουν το δρόμο για εξαιρετικά ε, σε σοβαρές παρεκκλήσεις. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή όπου πρέπει να γίνει σεβαστή η, η, σεβαστές οι προσδοκίες και να δημιουργηθεί με ένα πραγματικό δημοκρατικό ε, κράτος. Ε, τα δικαιώματα δε των κοπτών θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και να σταματήσουν οι διώξεις τους. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Είμαι blogger εδώ και πολλά χρόνια γιατί ε, το, το, το 1974 γλιτώσαμε από τους στρατιωτικούς τη δικτατορία για τη λογοκρισία και η εμπειρία μας μας έχει διδάξει ότι η πιο θεμελιώδης ελευθερία στην, σε περίοδους δημοκρατικής μετάβασης είναι η ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης οι προσωρινέ στρατιωτικέ αρχές. Αν δεν σέβονται αυτές τις θεμελιώδει ελευθερίε, όπως στην περίπτωση Αλ Αμπτελ Φατάχ, της γυναίκας του και άλλων, πάνω από 2.000 ε, ατόμων που έχουν προσαχθεί στα ε, στρατιωτικά του τελευταίου μήνε, αποδεικνύουν ότι αυτό που λαμβάνει η χώρα στην ε, Αίγυπτο είναι μία αδικία εις βάρος αυτών που έχασαν τη ζωή τους και αγωνίστηκαν εναντίον της δικτατορίας του Μουμπάρακ. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε, ξεκινώντας από την ύπατη ε, εκπρόσωπο, να ε, λάβουμε ε, τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να απαιτήσουμε το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών από τις ε, αρχές του, της Αιγύπτου και την απελευθέρωση αυτών των πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Våren 1848 svepte en våg av... ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άνοιξη είδαμε μια, ένα κύμα δημοκρατίας ε, να κινείται στην Ευρώπη το 1948 αλλά δεν νομίζω ότι η Αραβική Άνοιξη θα επικρατήσει κατά τον ίδιο τρόπο. Και για μας ε, ε, είναι αυτή η αποτυχία μία αποτυχία, είτε πρόκειται για στρατιωτική δύναμη ή δημοκρατική δύναμη. Ήταν η δική μας απόφαση. Αν είχαμε ζητήσει περισσότερο την ελευθερία με περισσότερους δικαστές, ε, μηχανικούς, η κοινωνία των πολιτών κλπ. θα είχαμε βοηθήσει πολύ καλύτερα το λαό εκεί. Έτσι ε, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε του λόγου για να μην έχουμε τι ίδιε αποτυχίε του kontekście. Για τρίτη φορά συζητάμε την κατάσταση στην Αίγυπτο. Κάθε φορά μέσα στα πλαίσια τη παραβία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την δίωξη των χριστιανών οποίος ε, ε, πέκρινε και κατέκρινε τις ε, Αιγυπτιακές αρχές. Το Σύνταγμα της Αιγύπτου εγγυάται την ελευθερία του πιστεύω ή του λόγου, αλλά το καθεστώς φέρεται σαν να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Φυλακίζουν bloggers, δημοσιογράφους, και εκπροσώπους οργανώσεων αντίθετους με την κατάσταση της στην Αίγυπτο. Επίσης διώκουν χριστιανούς. Η Αίγυπτος είναι εταίρος μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής γυτνίατσης ε, και θα θέλουν να πάρουν βοήθεια από μας. Θα πρέπει να τους πούμε ότι θα πάρουν τη βοήθεια αυτή μόνο υπό τον όρο να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Αιγυπτό για να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Για Ευχαριστώ, Η Αιγύπτος είναι ένα σημαντικός πολιτικός παράγοντας στην περιφερειακή ε, σταθερή δημοκρατική χώρα που σταθεροποιεί όλη την περιοχή. Ε, κάθε χώρα θα πρέπει να βρει το δικό της δρόμο προς τη δημοκρατία. Σωστό. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποια ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία του πιστεύω, της, του συνέρχεστε, του λόγου. Όλα αυτά είναι δικαιώματα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα για διαφορετικές ερμηνείες. Δηλαδή η απελευθέρωση ατόμων φυλακισμένων όπως τον Αμπτελ θα ήταν ένα δείγμα ότι η Αίγυπτο σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υποστηρίζω το πρώτο ψηφίσματο και θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει ούτως ώστε η Αίγυπτο να προχωρήσει προς την δημοκρατία, όχι μόνο προφορικά αλλά και στην πράξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τελευταίος ο κύριος Κάρας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε λίγα λεπτά ξεκινάω για ένα ε, συνέδριο στη Βηρητό και μετά θα πάω στην Αίγυπτο. Ακριβώς για το θέμα αυτό, ότι τα ψηφίσματα ε, και αυτά που άκουσα θα είναι η βάση των συζητήσεών μου. Είναι αυτονόητο αυτό. Η Αραβική Άνοιξη πέρασε. Η δημοκρατική άνοιξη όμως δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και χωρίς τη συζήτηση για την ε, ανοιξητρισκεία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς σύνταγμα πριν από τις εκλογές που να αναφέρεται στα δικαιώματα αυτά, δεν θα μπορούμε να είμαστε πιο τολμηροί για το μέλλον. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για τα ψηφίσματα αυτά που θα είναι πάρα πολύ σημαντικά στο ταξίδι μου και θα μπορούμε να πούμε για άλλη μια φορά χάρη των βασικών δικαιωμάτων ε, είναι η βάση όλων των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων όλων των φορέων όπου και να δρούν. Αυτό είναι ο δικό μας για ένα κράτος δικαίου και την δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, Ρε Πρόεδρος. Τώρα θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο σεβασμό των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ακρογωνία ο της τη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του γειτονέ τη. Το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο αναφέρει ότι οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο μέρη θα πρέπει να βασίζονται επί του σεβασμού των, των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά συμπεριλαμβάνουν ασφαλώς την ελευθερία ε, πίστης, ε, την ελευθερία του συνέρχεστε, ε, του ε, τους συνεταιρίζεστε και, τις και την ελευθερία έκφρασης. Εκ μέρους της Κομισιόν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η διεύρυνση και ε, η επαναδραστηριοποίηση ε, του νόμου έκταση κατάσταση, του καθεστώτος έκταση κατάσταση στην ε, Αίγυπτο μας ανησυχεί. Ιδιαίτερος μας ανησυχεί σε σχέση με την ελευθερία, με την ελευθερία έκφρασης, την λειτουργία της δικαιοσύνης και το δικαίωμα του συνέρχεστε. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί ασφαλώς η ε, τάξη, αλλά αυτά θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες ε, ατομικών δικαιωμάτων και πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται το πνεύμα ε, και οι προσδοκίες της Επανάστασης της 5 Ιανουαρίου καθώς επίσης και η επιθυμία των Αιγυπτίων πολιτών για δημοκρατικές εκλογές. Δυστυχώς η, Ευρωπαϊκή, ε, ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποσταλούν παρατηρητές για τις ε, εκλογές απορρίφθηκε από τις Αιγυπτιακές Αρχές. Θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παρέμβαση στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει συνδρομή ε, στις εκλογές μέσω της ε, κατάρτισης αρκετών ε, χιλιάδων παρατηρητών των εκλογών και βοήθεια προς την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή. Ο στρατιωτικός νόμος θα πρέπει να καταρριχθεί το συντομότερο δυνατό. Αυτή είναι η θέση της Ανώτατη τη ΥΠΑ της Εκπροσώπου και της Κομισιόν στο σύνολό της. Ε, υπό τον στρατιωτικό νόμο είναι δυνατή η φυλάκιση χωρίς δίκη αυτό ακριβώ ε, εφαρμόστηκε και στην περίπτωση του Αλά Απτελ Κατηγορείται ότι έχει υποκινήσει την βία κατά των στρατιωτικών αρχών και ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικό προσωπικό στις 9 Οκτωβρίου 2011. Ε, στρατιωτικές ε, δίκες πολιτών αρνούνται και καταργούν ένα τμήμα των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου στα πολιτικά δικαστήρια. Στις 15 Σεπτεμβρίου το Ανώτατο, δικαστήριο των, ε, το Ανώτατο Συμβούλιο των ε, Ενόπλων Δυνάμεων είχε υποσχεθεί ότι θα πάψει να δικάζει πολίτες σε, σε Αυτό όμως δεν ε, υλοποιήθηκε. η περίπτωση αλλά Φατάχ υπογραμμίζει την, την ε, το, την κρισιμότητα της κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει τις σοβαρές της ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ε, ενδεχόμενη ε, ερμηνεία των εξαιρέσεων με βάση τα, τις οποίες μπορούν να συνεχιστούν οι δίκες σε στρατοδικία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαμανάκη. Τελειώσαμε και με το θέμα της Αιγύπτου, ειδικότερα την περίπτωση του blogger Αλά Αμπτελ Φατάχ και μπορούμε να περάσουμε στις πιοφορίες. Καταρχήν θα ψηφίσουμε για, τα 6, για τις έξι προτάσεις ψηφίσματος για το Ιράν.